Καλησπέρα κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε. Βλέπω ότι έχουν μαζευτεί πολλοί εδώ στην αίθουσα και πολλά άτομα τα οποία συχνά δεν βλέπω ή, εν πάση περιπτώσει, δεν του ξέρω από εδώ, από την αίθουσα αυτή, από την επιτροπή αυτή. Αλλά να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη και στην έγκριση αυτή, στο σημείο 1. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσει. Ο κύριο Καμπ, Πρόεδρε, με έκπληξη είδα ότι αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε για το κατά πόσον η Επιτροπή ε, Μεταφορών θα κάνει ψήφισμα για κοινωνικά θέματα. Ξέρετε ότι στου συντονιστές, τη σχετική συνεδρία των συντονιστών, το συζητήσαμε επί το θέμα αυτό. Και η πλειοψηφία των συντονιστών θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει ξεχωριστό ψήφισμα για κοινωνικά τέτοια ζητήματα. Γιατί αυτό αποτελεί ουσιαστικά αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων. Ο συνάδελφο Ισμαλ Έρτουκ από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε ζήτησε να ψηφίσουμε παρόλα αυτά αύριο το πρωί και θεωρώ ότι είναι πραγματικά λυπηρό και υποβάλλω και ένσταση και σα ζητώ να το ψηφίσουμε ξεχωριστά αυτό αύριο το πρωί. Επαναλαμβάνω ότι εμεί ω ε, ΕΛΚ είμαστε υπέρ των κοινωνικών ζητημάτων ασφαλώ, αλλά σε συνάρτηση με τα θέματα που άπτονται των χερσαίων, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών και όχι σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα τη Επιτροπή Απασχόληση. Μάλιστα, λέει ο κύριο ε, Κράμερ, ζητήθηκε να αλλάξει η μερίσια καταξύ. Δεν υπάρχουν κανόνε ε, για τι επιτροπέ, αλλά ακολουθείται στο Κοινοβούλιο ένα γενικό κανόνα. Μπορεί φυσικά να γίνει έτοιμα για αλλαγή της ημερήσια διάταξης. Ο πρόεδρος ζητά να μιλήσει ένας υπέρ, ένας κατά και μετά θα ψηφιστεί η πρόταση αυτή. Αύριο, όχι σήμερα. Θέλει κάποιος να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. κυρία Φώστη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ βρισκόμουν στη συνάντηση πράγματι όταν έλαβε χώρα συζήτηση στους συντονιστές. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα που θίγει ο κύριος Βαντεκάμπ είναι σωστό. Εγώ στην Επιτροπή βρίσκομαι εδώ και πάνω από 11 χρόνια και φυσικά πάντα καλωσορίζουμε σχόλια και απόψεις συναδέλφων είτε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος είτε από την Επιτροπή Μεταφορών και συχνά ε, ε, τους δίνουμε και εμείς την άποψή μας, μας δίνουν αυτή τη δική τους. Αυτό που με ανησυχεί εδώ είναι το πεδίο αρμοδιοτήτων μας. Είναι πολύ σαφές εδώ στην Επιτροπή Μεταφόρων ε, αφορά ζητήματα μεταφορών. Παρότι υποστηρίζουμε τις θέσεις εργασίας ε, στις μεταφορές, γι' αυτό έχουμε μία δραστήρια Επιτροπή Απασχόλησης που ασχολείται με τα ζητήματα απασχόλησης. Γι' αυτούς τους λόγους πιστεύω η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να επανεστιάσει στο ποιε είναι οι προτεραιότητε τη. Είναι οι μεταφορέ, δηλαδή η μεταφορά ανθρώπων από το σημείο Α στο σημείο Β. Έχουμε τεράστιο φόρο εργασία για τη χρηματοδότηση, για ένα σωρό άλλα ζητήματα και πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, πιστεύω. Το ECR λοιπόν θα υποστηρίξει την άποψη που έθιξε ο κ. Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο κατά ο Ισμαήλ Ερτούχ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απορρίψετε αυτό το αίτημα. Το αίτημα αυτό δεν αποκρίνεται σε αυτά που συμφωνήθηκαν. Όλες οι αποφάσεις και συμφωνίες των συντονιστών έχουν έναν ε, χαρακτήρα συστάσεων, συστάσεων προς την Επιτροπή. Και η απόφαση αυτή η σε με πολύ ωριακή ψηφοφορία. Και γι' αυτό λοιπόν βγήκε και στην ατζέντα. Και πολύ λυπάμαι που ζητείτε να το ψηφίσουμε αυτό ξεχωριστά. Όταν κανείς είναι υπέρ των κοινωνικών ζητημάτων και θέλουμε και ένα περιβάλλον με ίσους όρους ανταγωνισμού, δεν υπάρχει λόγος να απορρίπτουμε ψηφοφορία τέτοιων ψηφισμάτων. Και χαίρομαι που τελικά τα τελευταία χρόνια καταλήξαμε στην ψηφοφορία των ψηφισμάτων. Τα διάφορα περιεχόμενα τα συμφωνήσαμε από πλευράς όλων των ε, ομάδων. Τώρα, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα με το συγκεκριμένο ψήφισμα, δεν μπορώ να πω. Με ξεπερνάει. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν έχει κάποιο σωστό στόχο αυτή, αυτό το αίτημα και γι' αυτό σας ζητώ να το απορρίψουμε. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Καταλήγουμε σε αυτά που είπαμε και στην προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι συντονιστέ, ε, ε, θα πρέπει να αποφασιστεί η Επιτροπή. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Έγκριση των πρακτικών τώρα, στο σημείο 2. Υπάρχουν ε, ε σημειώσει, ενστάσει. Τότε θα περάσουμε στο τρία, Συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την διαπραγματεύση σχετικά με τη Συμφωνία για τι Συναλλαγέ των Τομέα των Υπηρεσιών. ΤΙΣΑ. Ο Βιμ Κάμπ έχει το λόγο που είναι και εισηγητή και σα παρακαλώ όσοι εξέρχονται τι αιθούσει ήσυχα. Μην ενοχλείτε. Είμαι βέβαιο ότι θα μα καταλάβετε. Έχει το λόγο Βιμ. Πρόεδρε. Η οργανωμένη εκστρατεία του Ισμαήλ βγαίνει από την αίθουσα τώρα. Πολύ καλή δημοκρατική διαδικασία. Ε, δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα και αντίρρηση. Αλλά σήμερα το μεσημέρι θα μιλήσουμε για μια γνωμοδότηση την οποία η Επιτροπή Μεταφορών θα συντάξει για αυτή τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Πολύ σημαντική σύμβαση την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνάψει με 22 άλλες χώρες για το εμπόριο σε, στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Και αυτό ουσιαστικά ε, επηρεάζει όλους σχεδόν τις μεταφορές και σε κάθε περίπτωση την αυτιλία και την ε, αεροπορία τις μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές και κυρίως ε, τις, ε, την, ε, της παραδόσης δεμάτων, των deliveries. Υπάρχει λοιπόν μια διάσταση απόψεων. Μισό λεπτό διακόπτει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν γίνεται έτσι. Ε, τον Βιμ Φαντενκάμπ. Δική σου είναι Βιμ, αν εσυχάσουν, να συνεχίσεις. Δεν ε, καταλήξαμε στον ΚΑΤ να, καταλ... να πετύχουμε συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και 22 άλλες χώρες έλαβαν την πρωτοβουλία να συνάψουν μια ξεχωριστή σύμβαση. Και ξέρουμε όλοι ότι στην πολιτική δημόσια συζήτηση το TTIP είναι στο επίκεντρο της προσοχής, αλλά αυτή είναι μια πολύ πολύ σημαντική διαφορετική σύμβαση σε ό,τι αφορά Τη υπηρεσία. Έκανα λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότηση με τη βοήθεια των ε, υπαλλήλων, την οποία και θα καταθέσουμε προ την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και θα ήθελα να ζητήσω από του ε, συναδέλφου να μου πούν αν έχουν σχόλια για το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε και πού την ε, γνωμοδότηση αυτή. Ο Πρόεδρο, η Σκιωδή, η Καρολίνε Γκράσβαλτ Μάιντ. Ο Ισμαλ Έρτσουκ θα αναλάβει να μιλήσει εξ ονόματός τη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματο τη συναδέλφου η οποία δεν έχει καταφτάσει ακόμα γιατί ε, λόγω τη απεργία στα αεροπλάνα έχει κολλήσει στην κίνηση. Και θα ήθελα λοιπόν ε, να σα ε, αναφέρω τι είχε να σχολιάσει από πλευρά δική μου λοιπόν και τη κοιόδουση εισηγητρία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Κάμπ θεωρώ ότι αποτελεί μια καλή βάση η γνωμοδότηση, αυτή το σχέδιο γνωμοδότηση αυτή για τη μελλοντική διαπραγμάτευση. Να υποδείξω κάποια στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνει ακόμα η γνωμοδότηση. Για την ομάδα μα είναι πολύ σημαντικό η πρόσβαση σε διεθνεί συμβάσει να είναι στο μέλλον πιο κοινωνική και πιο διαφανή η προστασία του καταναλωτή του εργαζόμενου και κυρίως του περιβάλλοντος είναι στο επίκεντρο για μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών αλλοδαπή, από την αλλοδαπή θα πρέπει να τηρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκή Ένωση και τις λογικές συμβάσεις και τους κρατούς μισθούς. Τέτοιες λοιπόν ρυθμίσεις δεν μπορούν να θεωρούνται ως οικονομική επιβάρυνση αντιθέτως αποτελούν βασικά δικαιώματα και η γενική καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών, αποτελεί σύντημα καθοριστικό για την ομάδα μας, για την Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν απαιτούμε οι κοινοφελείς αυτές οι υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή. Επίσης, στο πλαίσιο ε, τροπολογίας θα υποδείξω και στον αρνητικό αντίκτυπο της ε, απελευθέρωσης υπηρεσιών στον τομέα της, ε, των υπηρεσιών αυτών. Και δεν θέλουμε λοιπόν να περάσουν τέτοια ζητήματα τα οποία έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την προάσπιση των προτύπων στον τομέα των αυτιλιακών μεταφορών και εδώ θα καταθέσουμε τροπολογίας και σε ό,τι αφορά τις οδικές ε, μεταφορές ε, και εδώ έχουμε να κάνουμε τροπολογίες και πέραν αυτών πρέπει να πω ότι προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία, σε μια επικοδομητική συνεργασία για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπατε πάρα πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Τάλτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου ε, του ECR θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ένα εξαιρετικό σχέδιο. Συμφωνούμε απολύτω με τον εισηγητή για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τη συμφωνία και υπογραμμίζει και την πολύ μεγάλη σημασία των μεταφορών στο παγκόσμιο εμπόριο. Έχουμε ένα αυξανόμενο ποσοστό εξάρτησης ε, στον τομέα αυτό και σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης χρειαζόμαστε πρόσβαση στις διάφορες αγορές του κόσμου όπου έχουμε το 90% των μελλοντικών προϊόντων. Πρόκειται για πολυμερή συμφωνία και ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι εντεταγμένη απολύτως ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ. Αλλά εδώ πρέπει να εστιαστούμε στην εναρμόνιση των κανόνων και, ε, και την άρση των εμποδίων το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 90% της ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης θα είναι στις υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε διαφανείς διαπραγματεύσεις για ισότιμο, κανόνε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού για όλους. Χρειαζόμαστε διασφάλιση για το μέλλον, διατηρώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας μην ξεχνούμε ότι τουλάχιστον στην οι μεταφορές στις ΗΠΑ έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά προστατευτισμού. Επομένως έχουμε μεγάλο αν θέλετε, διακύβευμα εδώ. Πρέπει να το προσέξουμε και στις αεροπορικές μεταφορές. Τώρα η ΤΙΣΑ είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να εστιαστούμε εδώ. Οι η θα είναι τεράστιες για μια επιτυχή συμφωνία για τη μελλοντική ευμάρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα εγώ θα είχα να υπογραμμίσω κάτι στις μεταφορές ε, στην οικονομία sharing ιδιαίτερα και ίσως επ' αυτού να κάνουμε μια πρώτη τροπολογία, αλλά γενικά συμφωνούμε απολύτως με τον εισηγητή. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Εμεί θεωρούμε τις διαπραγματεύσεις αυτές ως ε, πολύ σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι ολόψυχα στηρίζουμε το σχέδιο του κυρίου Βαντεκάμπ το οποίο καλύπτει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που έχουμε και ανησυχίες. Ο εισηγητής εστιάζει βεβαίως στα των μεταφορών και δεν πάμε στην κατεύθυνση που είχαμε πει πάει με την TTIP όπου καταψηφίστηκε παρότι δεν συζητούσαμε για θέματα μεταφορών. Αυτή η εστίαση είναι πολύ σωστή και μας δίνει τις κατάλληλες ευκαιρίες να έχουμε μια ευρύτατη, ευρύτατη στήριξη. Τώρα το άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η σημασία που δίνει ο εισηγητής στις θαλάσσιες μεταφορές. Είναι σημαντικό να προβλέπουμε κάποιους βασικούς κανόνες και να παρέχουμε ασφάλεια δικαίου στους Ευρωπαίους πλειοτήτες για την χρήση των λιμένων, τα δικαιώματα για τις ε, μεταφορικές συμφωνίες, αλλά κάτι που θα ήθελα να τονίσω εγώ και νομίζω ότι αποτυπώνεται ήδη στο προσχέδιο, είναι το καποτάζ. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως διαφανές το κείμενο. Πρέπει να άρουμε τα εμπόδια για το θαλάσσιο καποτέως και να ανοίξουμε την ε, αγορά αυτή. Γιατί σε κάποιες χώρες όπως γνωρίζουμε και η μεταφορά των άδειων ε, κοντέινερ μεταξύ δύο λιμένων δεν επιτρέπεται. Δηλαδή έχουμε ε, ένα υψηλό επίπεδο παράνοιας θα μπορούσα να πω μεταξύ κάποιων κανόνων που διέπνουν τα αγορά αυτή θα πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε την ε, διεθνή αλυσίδα οργάνωσης των μεταφορών. Αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις μας, ε, Πρόεδρε, αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε στήριξε ο πλευράς μας. Σας ευχαριστώ και βλέπω ότι κάποιοι είναι όρθιοι. Σας παρακαλώ, καθίστε. προκειμένου όλοι να μπορούν να ακούσουν και την ε, μετάφραση. Ο Φάμπιο Τεμάζη, επόμενο. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδέτηση. Δεν είναι μυστικό ότι η ομάδα των αριστερών, η GUNGL, είναι κατά τη ε, ΤΙΖΑ. Ε, Αυτό δεν είναι ευθύνη του εισηγητή, αλλά αυτών που αποφάσισαν να απελευθερέσουν περαιτέρω τον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Και μετά από όλε τι εμπειρίε που είχαμε στον τομέα των μεταφορών με την απελευθέρωση των υπηρεσιών ε, στην Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, κάποιοι άλλωστε μίλησαν και για θέματα διαφάνεια στι Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό που μέσω του Leaks ε, μάθαμε ότι πέντε χρόνια μόνο μετά τις διαπραγματεύσεις ε, θα δημοσιεύονταν τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων της ΤΙΖΑ και στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Ρουγουάη αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις πρόσφατα. Να τονίσω κάνα δύο θέματα παρόλα αυτά σε ό,τι αφορά τον ε, αρνητικό κατάλογο. Αυτό τι σημαίνει, ότι όλα όσα δεν ε, εξαιρούνται ρήτα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της ΤΙΖΑ. Και ε, πολύ φοβόμαστε ότι εδώ θα ισχύσει τελικά η αρχή της, ε, του πλέον ευνοούμενου, δηλαδή αν είναι ένα τομέα ο οποίο δεν εμπιπτεί στον τομέα εφαρμογή τη ΤΙΖΑ, αλλά είναι για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογή ε, τη ΣΕΤΑ, θα υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία και τα αρμόδια δικαστήρια. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι στον τομέα των μεταφορών ανησυχούμε ιδιαίτερα για θέματα τα οποία θάβονται εδώ στο Κοινοβούλιο, όπως η απελευθέρωση των χερσαίων μεταφορών. Και έτσι λοιπόν ακούσαμε από την πλατφόρμα Wikileaks υπάρχουν τα θέματα τα οποία γνωρίζετε και γι' αυτό λοιπόν θα επιμείνουμε στην τίζα να μην, να μην υπονομευθούν οι εργατικές ε, διατάξεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου και φίλου Βασικού που είναι εισηγητής ε, για το θέμα αυτό και που με ενημέρωσε για διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν μιλάμε για συμφωνία ε, τίθενται πολλά ερωτηματικά. Ερωτηματικά από αυτή τη στιγμή είναι το αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Εμείς λοιπόν ε, ως οικολόγοι Είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά αυτή την έκθεση. Οι προτάσει που κάνατε κύριε Βαντεκάμπ βρίσκονται ήδη στο ύψος των περιστάσεων, ικανοποιούν τον συναδελφό μου, αλλά εμείς θα θέλαμε να επισημαθεί περισσότερο η αρχή της αμοιβαιότητα, να ενισχυθεί στο σημείο ΙΙ της έκθεσή σας για να υπογραμμιστεί εντονότερα. Το δεύτερο είναι ότι η Συμφωνία της δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδυναμώσει τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική πτυχή, τον τομέα της ασφάλειας, αλλά και τον τομέα του περιβάλλοντος κυρίως. Εδώ μιλάμε για μεταφορές, αλλά πιστεύω ο στόχος είναι επίσης ε, να δίνουμε και μια εξήγηση όταν μιλάμε για μεταφορές. Μιλάμε για μεταφορές κυρίως εναέριες και θαλάσσιες. Αυτές πρέπει να αναφέρονται κύριος εδώ, οπότε είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι σημαντική η καχυποψία των καταναλωτών, των πολιτών, συγγνώμη, εν ώψη τέτοιων συμφωνιών, οπότε χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια. Ελπίζω λοιπόν κύριε Βαντεκάμπο ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα σημεία αυτά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, όχι πολλά. Εμείς ε, ευχόμαστε για τη συμφωνία αυτή να μην συνταχθεί έτσι όπως προχωράμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή με απόλυτη έλλειψη διαφάνειας. Και εδώ, όπως ακριβώς συνέβη και με την TTIP, ε, το Κοινοβούλιο δεν έδωσε καμία άποψη, δεν κλείθηκε να ε, δώσει κάποια άποψη. Μας ανησυχεί λοιπόν η εκπόνηση αυτής της συμφωνίας και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τις συμφωνίες του ΠΟΕ γενικότερα. Επιπλέον μας ανησυχούν επιπτώσεις για τις οδικές, θαλάσσιες, εναερίες αλλά και ταχυδρομικές μεταφορές και υπηρεσίες διότι θέλουμε να προστατεύεται το επίπεδο ποιότητας, να υπάρχουν κοινωνικές εγγύσεις, ανταγωνισμός και τα δικαιώματα των κρατών ε, για τις υπηρεσίες αυτής ε, κοινή ε, ωφελίας. Θέλουμε να αποκλειστούν δηλαδή οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος από τη Συμφωνία ΤΙΖΑ και θέλουμε να διατηρηθεί το δικαίωμα των κρατών να ρυθμίζουν την παροχή των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Επίσης θέλουμε να εισαχθεί μία ρήτρα ασφαλείας που θα βασίζεται σε προστατευτικά και προληπτικά σαφή μέτρα ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις κερδοσκοπίας και να διασφαλίσετε στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να υιοθετήσουν περιοριστικά δικαιώματα για την προστασία του γενικού συμφέροντος και του συμφέροντος των καταναλωτών. Επιθυμούμε λοιπόν προστασία των δεδομένων, ειδικότερα κατά την διαβίβασή τους σε τρίτες χώρες. Αυτές είναι οι ανησυχίε που μα απασχολούν κυρίως εμά και ελπίζουμε ότι εφόσον εγκριθούν οι δικές μας τροπολογίες, θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ευρία βάση επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μαρή Χριστίνα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι. Διαβάζοντας αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση που συζητάμε σήμερα, συνάγω ένα σαφές συμπεράσμα που δεν θα σας εκπλήξει θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναδούμε ολόκληρη τη γνωμοδότηση και σας προτείνω να την αντικαταστήσουμε να αντικαταστήσουμε την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού που καλεί την Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου να την αντικαταστήσουμε ως, με την εξή φράση το Κοινοβούλιο ζητά από την Κομισιόν να αποσυρθεί αμέσως από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ΤΙΣΑ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πολλοί από σας έχουν πει οι διαπραγματεύσεις αυτές ξεκίνησαν με απόλυτη αδιαφάνεια. Χρειάστηκαν ε, στοιχεία και αποκαλύψει από την Wikileaks πέρυσι ε, για να μάθουν οι πολίτες μας κάποιο μέρος του περιεχομένου. Τα όσα μάθαμε ήταν τόσο επικοδομητικά που δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί πολλοί από τους λαούς μας αφέθηκαν στην άγνοια. Και για μας αυτό δεν μεταφράζεται σε δημοκρατία. Στόχος της Κομισιόν είναι πολύ είναι κάτι πολύ σαφές να άρει τα τελευταία τελωνιακά ε, εμπόδια για να ενθαρρύνει τον φιλελευθερισμό. Εξάλλου υπόθηκε ο σημερινός κόσμος δεν γνωρίζει πλέον σύνορα. Ταυτόχρονα ορισμένες ε, χώρες αναφέρεται ότι δυστυχώς αντιτίθενται στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Κύριε γιατί το ίδιο σκέφτεστε και εσείς όταν λέτε ότι η Κομισιόν πρέπει να δράξει την ευκαιρία να ενοποιήσει τις σημερινές νομοθεσίες και πρακτικές όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές σε ένα διεθνές κείμενο ε, νομικά ε, δεσμευτικό το οποίο θα ανοίξει το δρόμο σε περαιτέρω ε, ε, μέτρα προστατευτισμού από τα μέρη. Ποιο μα έδωσε δικαίωμα να αποφασίζουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθο στη θέση των λαών μα. Αν αύριο δηλαδή οι Γάλλοι αποφάσιζαν ή επιθυμούσαν να αποκαταστήσουν το δημόσιο μονοπόλιο των αυτοκινητοδρόμων, αυτό θα ήταν αδύνατον επειδή θα υπήρχε μια τέτοια συμφωνία σαν αυτή. Το ίδιο ισχύει για όλε τι υπηρεσίε που δεν θα έχουν εξαιρεθεί κατά την υπογραφή τη συμφωνία. Είτε μιλάμε λοιπόν για το τοπικό, το περιφερειακό, είτε για το εθνικό επίπεδο, οι λαοί θα δυνατούν συνεπώς να επαναφέρουν ε, οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση ή ε, απελευθέρωση και το μόνο που θα μπορούν να κάνουν θα είναι να προχωρήσουν σε περαιτέρω ε, απελευθέρωση. Τέλος, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν να πούν κάτι για τα διάφορα κεφάλαια στον τομέα όμω των μεταφοράνων υπάρχουν διαφορετικέ απόψει μεταξύ των κρατών μελών. Αν η Γαλλία λοιπόν επιθυμούσε οι σιδηρόδρομοι να παραμείνουν δημόσιο μονοπόλιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει το αντίθετο και αποφασίσει ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών οι σιδηρόδρομοι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν και να του ανοίξουν στον ανταγωνισμό ε, χώριο και ξένο, ε, εκεί φυσικά η Γαλλία δεν θα μπορεί να αντιτεθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ υπερασπίζομαι εγώ τα συμφέροντα των Γάλλων και δεν εξυπηρετώ ε, δημοκρατικά συμφέροντα δίθεν όσων υπερασπίζονται ένα κόσμο χωρίς σύνορα. Οπότε επιμένω η Επιτροπή μας να ζητήσει, να σταματήσει άμεσα αυτή η διαπραγμάτευση εξ ονόματος της εθνικής κυριαρχίας και της ελευθερίας των λαών. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΑΕΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιο άλλο εδώ. Πείτε μα και ποιο είστε. Σωστά κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Λίτζι Πόλη από τη Γενική Διεθνή Εμπορίου. Ασχολούμαι με τις υπηρεσίες και με τη Συμφωνία ΤΙΣΑ. Επίσης, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τη συζήτηση αυτή και γενικά τα υποστηρικτικά λόγια που ακούστηκαν εδώ για τη διαπραγματεύση αυτή η οποία όπως υπόθηκε είναι πολύ σημαντική διότι οι υπηρεσίες μεταφορών ε, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25% της συνολικής αξίας των υπηρεσιών και ειδικότερα ανέφεραν ε, μερικά μέλη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές ε, είναι εξαιρετικά σημαντικές ως τρόπους μεταφοράς μεταφέρουν πάνω από το 90% των εμπορευμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς λοιπόν προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από την αποτυχία της συνέχισης ε, της ε, συμφωνίας GATT ε, και της DDA είναι η πρώτη αυτή λοιπόν προσπάθεια να προχωρήσουν κάπως οι εργασίες που είχαν ξεκινήσει στη, με τη Γενική Συμφωνία ε, Εμπορίου και Υπηρεσιών, την ΚΑΤ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα πολλά σχόλια που ακούστηκαν, ειδικότερα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, γιατί άκουσα κάποια σχολεία περί διαφάνειας. Η διαπραγματεύση αυτή πιστεύω είναι υπόθυγμα διαφάνειας θα έλεγα όλα τα έγγραφα τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση με την παρακολούθηση αλλαγών, με όλα τα σχόλια των διαφόρων χωρών που βρίσκονται γύρω από το τραπέζι, όλα αυτά τα στοιχεία είναι στη διάθεση της Επιτροπής αυτή. Έχουν διαβιβαστεί στα κράτη-μέλη, έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Ε, είναι λοιπόν στη διάθεση όλων των Ευρωβουλευτών ε, αν θέλουν να ρίξουν μια ματιά. Όχι μόνο δηλαδή στα τελευταία κείμενα που απορρέουν από κάποιε συζητήσει, που φυσικά δεν υπάρχουν ακόμα γιατί οι συζητήσει ακόμα συνεχίζονται, αλλά σε όλα τα στάδια των συζητήσεων. Αυτά είναι λοιπόν το πρώτο μου σχόλιο όσον αφορά τη διαφάνεια και νομίζω ότι η κυρία Ρέντιν νομίζω ε, επένεσε τις διαπραγματεύσεις μάλιστα της ε, από αυτή την απόψη. Ε, ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Όλοι γνωρίζουμε φυσικά ότι στις μεταφορές είναι σημαντικές οι δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης των, του επίπεδου ποιότητας ούτε ύπαρξης άλλων προβλημάτων που να σχετίζονται με κοινωνικά θέματα. Ε, όπως τα προστατεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί το λέω αυτό, διότι ε, διαπραγματευόμαστε βάσει συνένεσης πρώτα απ' όλα, αλλά όπως και σε άλλες διαπραγματεύσεις και στη Δύση έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε επιφυλάξεις, που είναι επιφυλάξεις όπως λέει ο λόγος, όπου προστατεύουμε κάποιους τομείς όπου παραδοσιακά είχαμε επιφυλάξει όπως για δημόσιες υπηρεσίες ε, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων μεταφορών. Οπότε εδώ θα ήθελα να διασκεδάσω τις ανησυχίες ε, που ακούσαμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο πάλι όχι εσείς, ο Βίμπτον Νεκάμπ. Πρόεδρε, πολύ ευχαριστώ να ευχαριστήσω και όλους τους κοιόδης εισηγητές για τις παρατηρήσεις που έκανα. Αλλά ανησυχώ κάπως. Συμφωνώ πολύ με τους, ε, τον συνάδελφο από την Να προσέξουμε, η γνωμοδότηση των ε, μεταφορών να μην επιβαρυνθεί με διάφορες γενικόλογε παρατηρήσει για την εμπορική πολιτική, για το τι. για κάθε είδους πρόβλημα το οποίο μπορεί κανείς να θεωρεί ότι υπάρχει. Καταλαβαίνω τις παρατηρήσει των συναντέλφων από την Κούρ, αλλά αν θέλουμε να τα βάλουμε τώρα όλα αυτά μέσα στην γνωμοδότηση, δεν θα είναι πλέον γνωμοδότηση από την Επιτροπή μεταφορών. Και αυτό είναι το μεγάλο δίλημα ενώπιον του οποίου βρίσκομαι. Η ε, ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκός ε, κλάδος των μεταφορών θα ωφεληστεί από τη σύμβαση αυτή. Θα μας ανοίξει πάρα πολλές ευκαιρίες και στις αεροπορικές μεταφορές και στις χερσαίες μεταφορές. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και δεν νομίζω ότι στη γνωμοδότησή μου θα πρέπει να βάλω κάθε είδους γενικά εμπορικά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένω να αναφερθούν. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι για την 3η 24 Νοεμβρίου στις 9.30 ε, έχουμε προγραμματίσει συνάντηση των ε, σκιωδών. Ελπίζω να έχω λάβει τις ε, τροπολογίες σας, γιατί η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα ψηφίσει στις 10 Δεκεμβρίου, άρα θα πρέπει να βιαστούμε κι εμεί, Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήθελα με την βοήθεια της γραμματεία να φροντίσουμε να ψηφίσουμε 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή μας. Και ασφαλώς και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλια που έκανε και σε ό,τι αφορά θέματα διαφάνεια, θα πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά όπως σας είπα, δεν μπορούμε να ε, κάνουμε μια σύμβαση, να διαπραγματευτούμε μια σύμβαση με 751 άτομα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να κάνω μια παρατήρηση για το τελευταίο αυτό ζήτημα. Ως ε, Επιτροπή έχουμε ασφαλώς ε, δικαίωμα να κάνουμε τροπολογίες. Το τι γίνεται τελικά στην ψηφοφορία το είδαμε στο TTIP γιατί κάποιοι, κάποιες ομάδες και κάποιε επιτροπέ ε, που δεν του άρεσε κάποια τροπολογία, τελικά την ψήφισαν στο τέλο. Και εμεί ε, ήμασταν οι μόνοι που δεν επεκταθήκαμε στο θέμα αυτό. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση προ όλου μα. Για να πετύχουμε τελικά ένα ψήφισμα το οποίο θα μα επιτρέψει να μπούμε στη συζήτηση και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 12 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Είναι λίγο ωριακά τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε και επιλογή τι να κάνουμε. Και τώρα να περάσουμε στο 4 της ημερίας της διάταξης προς μία πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η Μέρια Κίλονεν είναι η συγκήτρια, της δίνω πάρα αυτό το λόγο. Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν με μεγάλη χαρά που συνεργάστηκα με όλους επί της ε, γνωμοδότηση αυτή ε, για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Συνολικά, λάβαμε διάφορες προτάσεις ε, τροπολογιών που δείχνουν ότι η Επιτροπή Τραν έχει μια αρκετά ενιαία άποψη επί της ψηφιοποίησης και επί των ανησυχιών και κινδύνων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή βιομηχανία τουρισμού και μεταφορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για μια πολύ επικοδομητική συνεργασία. Οι συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, θα ψηφιστούν αύριο και θα ήθελα επ' αυτών να πω δύο λόγια. Καταρχάς ε, η Επιτροπή επί των συμβαστικών προτάσεων θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η εργασία έχει αλλάξει μέσω της ε, ψηφιοποίησης και επομένως πρέπει να ενισχυθεί η κατάρτιση των εργαζομένων ώστε να επικαιροποιούνται οι δεξιότητές τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ε, του ψηφιακού χώρου και της ε, τεχνολογίας. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουμε ότι ανταποκρινόμαστε προς τις προσδοκίες των χρηστών. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιη ότι χωρίς τις ψηφιακές ευκαιρίες που μας ανοίγονται αυτή τη στιγμή μπορούμε να τα επιτύχουμε αυτό. Τουλάχιστον όταν μιλούμε για τις αλυσίδες που ασχολούνται με τις μεταφορές και την κινητικότητα και τις δυνατότητες που έχει ο κάθε χρήστης. Υπό την οπτική λοιπόν γωνία του χρήστη χρειαζόμαστε πολυεπίπεδα κέντρα πληροφοριών, έκδοση εισιτηρίων και είναι απορίας άξιο ότι κινούμαστε προς το 2016 και είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται να σκάψουμε ένα τούνελ μέσα σε ένα βουνό παρά να εκδώσουμε ένα εισιτήριο που να συνδυάζει διάφορα μέσα μεταφορών. Η ψηφιοποίηση φέρνει μαζί της διάφορες προκλήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, Και πλέον δεν πρέπει να μιλούμε απλώς για υποδομές υπό την έννοια των μεταφορών υποδομών, αλλά καθότι οι ψηφιακέ υπηρεσίε γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς και απαραίτητες, θα πρέπει να έχουμε επαρκή ικανότητα μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων. Και τα διάφορα λόγια που έχουν ακουστεί και οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί δεν έχουν όλα αυτά συμπεριληφθεί σε όλες τις συμβαστικές προτάσεις, όμως προσπαθήσαμε να έχουμε μια σαφή δέσμη προτάσεων που να μπορούμε να την υποβάλλουμε ως κοινή έκθεση, ως συνενετική κοινή έκθεση με τις βασικές στοιχείες των μεταφορών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Σας ευχαριστώ. Η επόμενη Ευχαριστώ, Πρόεδρε, η κυρία θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον, ε, την εισηγήτρια για την ε, εργασία της. Ε, νομίζω ότι κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα πλέον σε μια θέση την οποία θα ψηφίσουμε αύριο για να παρουσιάσουμε προς την Επιτροπή ΙΤΡΕ και Επιτροπή ΙΝΚΟ. Όπως είπε λοιπόν η εισηγήτρια, είναι τεράστια το δυναμικό του τομέα αυτού για την ε, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και όλου του τομέα της επιμελητίας των ηλεκτρονικών συνόρων, των τελωνίων. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι ακόμα έχουμε τέτοια χαρτούρα στα σύνορα και η εισαγωγή ηλεκτρονικών και ψηφιακών συστημάτων θα βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση και τη, τις και το εμπόριο και ασφαλώς την κοινωνική οικονομία, τον τομέα του τουρισμού. Είναι πολύ σημαντική η ψηφιοποίηση και στο πλαίσιο αυτό. Όπως είπε λοιπόν η συγκήτρια, θα πρέπει να εκπαιδευτούν και όλοι όσοι θα εργαστούν στον κλάδο αυτό. Καλώς ορίζουμε λοιπόν όσα είπε η συγκήτρια και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στην διατύπωσή μας, να επικεντρωθούμε στα θέματα που άπτονται ε, κυρίως στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού. Ευχαριστώ και θα δούμε τι θα γίνει αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του και κυρίω για την προσέγγιση του. Ε, το ανοιχτό μυαλό με το οποίο αντιμετώπισε όλους τους ε, σκιώδεις συζητητέ. Ως ε, εγώ σκιώδης εισηγήτρια, εγώ εισηγήτρια έχω να πω ότι υποστηρίζουμε όλες τις προτάσεις συμβιβασμού. Αντιμετωπίζονται εδώ όλες οι διαδικασίες ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς των μεταφορών και υποστηρίζουμε επίσης και την πρόταση των έξυπνων συστημάτων στις μεταφορές. Επίσης είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η γνωμοδότηση περιλαμβάνει και την πτυχή της ε, προσβασιμότητας ε, ε, ηλικιωμένων ατόμων στα ψηφιακά συστήματα. Δεν πρέπει να αποκλείεται αυτή η ηλικιακή ομάδα από την ψηφιοποίηση. Δεν μπορεί η ψηφιοποίηση να αποτελεί εμπόδιο για ηλικιωμένου ή για άλλε ευάλωτε ομάδε. Επίση, υποστηρίζω την άποψη ε, τη εισηγήτρια ότι πρέπει να διασφαλίζεται η κατάρτιση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης. Στο τομέα των μεταφορών και του τουρισμού θα θέλαμε να μην υπάρχει γεωγραφικός αποκλεισμό όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσπελασμένες παντού, όπου και να βρίσκεται κανείς. Είμαι πεπισμένη ότι όλοι θα στηρίξουν αύριο στην ψηφοφορία αυτή τη γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια και της εύχομαι ε, καλή επιτυχία και ελπίζω ότι πολλές από ε, τις πτυχέ που ανέφερα θα συμπεριληφθούν ε, στην έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, η διερμηνία έρχεται λίγο πιο μετά από την αρχική ομιλία. Ο κύριος Ντάλτον έχει το λόγο τώρα. Um, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ το καλύπτω αυτό στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και επομένως μιλώ και υπό την ιδιότητα αυτή. Εδώ έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές για όλους τους κλάδους και θα αλλάξει και τις μεταφορές όπως, και την, ε, όπως άλλαξε και η γεωργία με τη βιομηχανική επανάσταση, με, τους, ε, με την ατμομηχανή, τους ιδεοδρόμους. Η ψηφιακή οικονομία θα κάνει αντίστοιχες αλλαγές θα επιφέρει. Τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με αρκετέ από τις συμβαστικέ προτάσεις που έχουν υποβληθεί για τις ε, πλατφόρμες, για τη συνεργατική οικονομία, για, τα, για την έκδοση εισιτηρίων ε, πολυμέσων, πολυμεσικών, πολυτροπικών. Και έχουμε εδώ τεράστιες δυνατότητες για τις αεροπορικές μεταφορές. Γιατί χωρίς πρόσθετο κόστος θα προσφέρει τεράστια αύξηση συνδυάζοντας τη ζήτηση με την προσφορά και νομίζω ότι όλες οι χώρες σε αυτό θα έπρεπε να εστιάζονται. Αυτά είναι πολύ θετικό ότι έχουν επισημανθεί και τα στηρίζουμε. Αλλά μία, μία παρατήρηση για λίγο προσοχή, όπως η πρόταση έχει αυτή τη στιγμή, ίσως υπογραμμίζει υπερβολικά την επικουρικότητα όταν μιλούμε για τα φορολογικά, τις εργασιακές συνθήκες και την προστασία των καταναλωτών. Αυτά είναι εθνικά θέματα. Και στην Επιτροπή εσωτερική Αγοράς αναγνωρίζουμε ότι είναι εθνικής Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θίγουμε αυτά τα θέματα. Ο κύριος Τελίτσκα. thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν το λέω λόγω ευγένεια και παράδοση, αλλά πραγματικά ευχαριστώ την εισηγήτρια και εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι δικές μας προτάσει και οι περισσότερες προτάσει έχουν ληφθεί υπόψη στις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή γνωμοδότηση και οι συμβαστικές λύσεις ε, προσφέρουν μια συνολική ισορροπία και για τις μεταφορές και για τον τουρισμό. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλά ισορροπημένη λοιπόν προσέγγιση και για τις επενδύσεις και για τις υποδομές και για τους εργαζομένους, την κατάρτιση και τα δικαιώματα των επιβατών. Πολλά έχουμε πει για την ψηφιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό για τον κλάδο αυτό όπως και για πολλούς άλλους και ελπίζω πραγματικά ότι αυτό το input θα μπορέσει να βοηθήσει να μπορέσουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα σύστημα μεταφορών άξιο του 21ου αιώνα. Όπως υπογράμμισαν και άλλοι επειδή δεν θα επαναλάβω η ψηφιοποίηση των, ε, του συστήματος μεταφορών και τουρισμού θα οδηγήσει σε νέες τάσεις και συμπεριφορές από πλευράς των καταναλωτών και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα βήματα που θα χρειαστούν για τις απαραίτητες υποδομές και θα χρειαστούμε και το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει χωρίς την απαραίτητη αξιολόγηση αντικτύπου. Και αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να το υπογραμμίσω. Επίσης, θα έλεγα ότι εκτιμώ ιδιαίτερα ότι σε αντίθεση με άλλες επιτροπές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ καλά τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά πλαίσια, τους πόρους για τα των μεταφορών και του τουρισμού και πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διείσδυση των μεταφορών και της ψηφιοποίηση, αλλά βέβαια δεν έχουμε δυστυχώς τα ίδια μέσα στη διάθεσή μας όπως άλλες επιτροπές, όπως η Γιούρη. Παρόλα αυτά, είναι ένα, ένα σχόλιο παρένθεση ο πλευράς μου, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνουμε να εκφράσουμε μια ευρύτατη συνένεση στις γνωμοδοτήσεις μας. Εν πάση περιπτώσει εκτιμώ απολύτως την πρόταση αυτή και θα την υποστηρίξουμε με χαρά. Τώρα τις ε, τροπολογίες ε, χωριστής ψήφου που δεν ασχολούνται με τα μεταφορικά και του τουρισμού δεν θα θέλαμε να τις υπερψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ πάνω να συγχαρώ τη συναδέλφο και η εισηγήτρια για τις προσπάθειες της. Οι συνεδριάσεις για την εξέβραση συμβιβασμών χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη συλλογική ευφυΐα και μεγάλη ευχαρίστηση θα μπορούσε να πει κανείς. Πραγματική ευχαρίστηση. Η γνωμοδότηση αυτή πιστεύω είναι ουσιώδου σημασία. Γιατί διότι η γνωμοδότηση αυτή δείχνει ότι ο ψηφιακός κόσμος ε, θα δώσει μια νέα μορφή στην κινητικότητά μας αλλά θα δημιουργήσει και νέες μορφές οικονομίας και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε διότι η τεχνολογία καλό είναι να ενταχθεί στην αστική κινητικότητα μπορώ εγώ να σας το πω από πρώτο αλλά οι συμπεριφορές αλλάζουν. Ειδικότερα με τους τομείς αυτούς, ε, τους κλάδους αυτούς που όλο και περισσότερο ε, αμφισβητούν τις καινοτομίες, ε, τη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, κοινών αυτοκινήτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να ψηφίσετε την τροπολογία μου 46 αύριο διότι στον ψηφιακό χώρο αυτή τη στιγμή υπάρχει η επιχείρηση Uber. Αν θεωρήσουμε ότι Uber είναι ένα καθαρό ε, παράδειγμα επανάστασης της συνεργατικής ε, αυτής της οικονομίας, ε, θα ήταν επικίνδυνο να θεωρήσουμε ότι η Uber είναι αυτό που προωθεί η ίδια ως εικόνα δική της μια ψηφιακή υπηρεσία. Η Uber παραμένει μια επιχείρηση που επηρεάζει σημαντικά τις αστικές μεταφορές σε πολλά κράτη-μέλη και η αλήθεια είναι ότι παρέχει καλές υπηρεσίες αλλά μην ξεχνάμε τι προβλήματα θέτουν αυτές οι υπηρεσίες προβλήματα σε θέματα ασφάλειας ε, έλλειψης κοινωνικής προστασίας ε, ασφάλισης η τροπολογία λοιπόν αυτή είναι σημαντική διότι οι απαντήσεις που δίνονται σήμερα σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα ε, είναι διαφορετικές ε, ε, από κράτος σε κράτος και από πόλη σε πόλη μάλιστα. Η, με την τροπολογία μου λοιπόν ενθαρρύνω την ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου σε θέματα ανταγωνισμού, ελάχιστων κοινωνικών απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούνται. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο, δεν μπορούμε να πούμε είμαστε κατά. Πρέπει να αρχίσουμε να ρυθμίζουμε χωρίς να πνίξουμε την κοινοτομία ε, καινοτομία που θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη ε, στο μέλλον για την οικονομία ε, και που επιθυμούμε να υπάρχει υπό σωστέ συνθήκες όμως για αυτό το λόγο πιστεύω βέβαια ότι, παρόλα αυτά πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά καλή και οι οικολόγοι θα ψηφίσουν υπέρ ευχαριστούμε κύριε Λόντγκρεν ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λοιπόν Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξαιρετική δουλειά του εισηγητή και συμφωνώ απολύτως με την κυρία Ντελή επί του Uber. Πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα ταξί. Αλλά υπό την έννοια την ψηφιακή έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Είναι ένα αεραστεχνικό σύστημα, όπως λέει η κυρία Ντελή, όπου οι επιβάτες έχουν κίνδυνο Υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, έλλειψη ελέγχων, έλλειψη ελέγχων και φορολογικών. Πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα που επιχειρεί να καταστρέψει, να διασπάσει την αγορά των ταξί. Και υποστηρίζουμε την πρόταση κυρία Ντελή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Μαρή Κριστίνα Γιούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλούμε για την ε, προτεραιότητα υπαριθμών 2 της Κομισιόν Juncker. Η ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό το χαιρετίζει η συγκεκριτρία, εγώ όχι. Και εκεί θέλουμε να άρουμε όλα τα συνοριακά εμπόδια. Συζητούμε δηλαδή επί των ψηφιακών, παρακάμπτοντας για μία ακόμα φορά την αρμοδία των κρατών μελών. Οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει αντιθέτω, αποσκοπούν στην επιστροφή της πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη ώστε να είναι ελεύθερα να επιλέξουν μια κοινωνία ελεύθερων ψηφιακών συναλλαγών χωρίς ελέγχους ή μια κοινωνία που θα επιχειρεί να προστατεύσει, να τα προσωπικά δεδομένα των συμπολιτών τους. Υπό την έννοια της ε, οικονομικής ε, ανάπτυξης Είμαστε πλέον σε μια ροπή άναρχης χρήσης των ψηφιακών μέσων. Ε, έχουμε μια ψηφιακή απικιοποίηση η οποία επιτρέπει στις μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Google και η Facebook να γνωρίζουν όλες μας τις μετακινήσεις, τις συνήθειές μας, τον τρόπο ζωής, τα έξοδά μας και πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο, θα γνωρίζετε ότι κάποιοι εξαιρετικά καταρτισμένοι προγραμματιστές απεκάλυψαν την κατασκοπία αυτά, την κατασκοπία που συμβαίνει κατά των πολιτών από την Microsoft μέσω του Windows 10 και αυτό πλήττει και τους καινούριου υπολογιστές και τους παλαιούς γιατί πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε συνέχεια αναβαθμίσεις λογισμικού. Λογισμικού που απορροφά όλα τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Επομένως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θεμελιώδες, θεμελιακό ζήτημα που είναι η προστασία της ελευθερίας και της ιδιωτικής ζωής. Που και αυτές οι αρχές πρέπει να εκφράζονται από την Επιτροπή μας. Τώρα, δεν είμαι σε καμία περίπτωση εχθρική και δεν είμαστε εχθρικοί προς τα ψηφιακά μέσα. Αντίθετα, είμαστε πεπισμένοι ότι έχουν πολυάριθμα πλέον εκτήματα για την καλύτερη διαχείριση των ροών πλοήγησης, για παράδειγμα, ή μετακίνησης. Αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα επιλύσει όλα μας τα προβλήματα. Δεν πρόκειται για κάποιο μαγικό ραβδί κατά της ε, επιμόλυνσης, ε, κατά του κυκλοφοριακού των προβλημάτων που έχουμε. Αναφερθήκατε στο Uber. Δεν είναι παρά η συνέπεια και το αποτέλεσμα των πολιτικών τις οποίες υποστηρίζετε και εξακολουθείτε να υποστηρίζετε της απόλυτης ε, φιλελεύθερης ανταλλαγής υπηρεσιών και εμπορίου. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τη κατάλληλη θέση της ψηφιακής ε, τεχνολογίας στη ζωή μας και επιμένω ότι η προστασία των νομικών ελευθεριών και, της, ε, και του ιδιωτικού βίου θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Επιμένω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιζαμπέλ Ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το κείμενο αυτό το οποίο με βρίσκει σύμφωνη. Εκτιμώ ιδιαίτερα και τη συνεργασία των σκιωδών για την επιτευχή των συμβιβαστικών. Ήθελα να πω ότι η ενιαία αγορά έχει σκοπό την άρση των εμποδίων για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης. Μιλάμε για διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και τα λοιπά, οπότε είναι ε, αγαθό να σκέφτεται κανείς ότι δεν υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Τα στοιχεία λοιπόν να χρησιμοποιούνται και αυτή τη χρήση εμείς μπορούμε να τη ρυθμίσουμε, όχι να την απαγορεύσουμε, για την προστασία των πολιτών. Ε, σίγουρα απαιτείται εξυγχρονισμός ε, του ρυθμιστικού πλαισίου για τον νέο ψηφιακό κόσμο και αυτό αφορά τις μεταφορές ε, και τον τουρισμό φυσικά αφού η Επιτροπή μας ονομάζεται Μεταφορών και Τουρισμού και έτσι έχουμε προετοιμάσει ένα κείμενο πρωτοβουλίας ε, για τον τομέα του τουρισμού για το μέλλον που αφορά τα ζητήματα και της ψηφιοποίησης και το ζήτημα της συνεργατικής οικονομίας. Υπάρχει περίπτωση να πέσουμε στην παγίδα να δαιμονοποιήσουμε οι υπηρεσίε αυτέ που υπάρχουν εδώ και χρόνια, όπω και η ψηφιοποίηση, και που σε ορισμένε περιπτώσεις ε, έχουν ε, αποδειχθεί επικοδομητικές ε, στις μεταφορές και στον τουρισμό. Δεν πρέπει λοιπόν να εμποδίζουμε, πρέπει να επιτρέψουμε οι δραστηριότητες, ειδικότερα οι εικονικές δραστηριότητες, να διεξάγονται μεν, αλλά μέσω κάποιας ρύθμισης που ακριβώς όπως υπογραμμιστήκε προηγουμένω να μην καταπνιγεί μια οικονομική δραστηριότητα. Αναμφίβολα η καινοτομία ανέκαθεν δημιουργούσε μείωση των θέσεων εργασίας. Αυτό όμως ε, δεν αποκλείει ε, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της δημιουργίας νέων υπηρεσιών και μεγάλων μάλιστα οικονομικών δραστηριοτήτων και σε αυτού του τομεί. Ευχαριστούμε πολύ. Στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουμε τώρα το λόγο. Βον Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει πώς η ενιαία ψηφιακή αγορά περνάει από την ψηφιοποίηση πολλών πολλών τομέων και πολλών πτυχών. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την συζήτηση αυτή και στην ένταση της και την ποιότητα της συζήτησης της ιστορικής που έχει γίνει. Καλωσορίζουμε συνολικά την γνωμοδότησή σας και την σχετική συζήτηση που έγινε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία λόγω της ε, ευρεία εφαρμογή της ψηφιοποίηση ενδεχομένω να σα οδηγήσουν σε συγκεκριμένε ε, συστάσει, σε συγκεκριμένες... Ε, παρατηρήσεις ε, που θα θέλατε να βάλετε στην χρηματοδότηση και θα δώσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση μου. Μάλιστα, και εγώ αυτό πρότεινα. Η κυρία Κλέρ Ντεπρέ από την Γενική Διεύθυνση μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια για να πω ότι και εμείς από την πλευρά της DG Move καλωσορίζουμε φυσικά αυτή την γνωμοδότηση για να αντιδράσω στη συζήτηση που έγινε. Η ψηφιοποίηση τη μεταφορές δεν είναι κανόνα ε, που πρέπει να υπάρχει έτσι, ε, από μόνο του. Ε, βοηθά στην αποτελεσματικότητα, στην πολυτροπικότητα των μεταφορών, στην αξιοποίηση της αλλαγής των συμπεριφορών, στην προσφορά νέων δυνατοτήτων χάρη στα ψηφιακά συστήματα και το δίνει περισσότερη προσοχή στους επιβάτες ε, ε, και μάλιστα σε ε, ανθρώπους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με προβλήματα κινητικότητας και ούτω καθεξής. Όσον αφορά μία από τις τροπολογίες που συζητήσαμε, όπως ξέρετε, εμείς από πλευράς Κομισιόν υποστηρίζουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα εφόσον πληρούνται απαιτήσει ασφαλείας, φορολογικές, κοινωνικού χαρακτήρα που έχουν ε, θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Κάτι για τα εισιτήρια. Αναφέρατε πολλά για τα εισιτήρια, για την έκδοση εισιτηρίων και σε κάποιες τροπολογίες αναφερθήκατε και στα δικαιώματα των επιβατών. Το έχω ξαναπεί παλιότερα. Να έχουμε πρώτα απ' όλα ίσως σωστές πολυτροπικές πληροφορίες ώστε όταν περνάμε στην έκδοση εισιτήριων και στα δικαιώματα των επιβατών να έχει προλυνθεί το έδαφος να είναι έτοιμα τα πράγματα για την προστασία των επιβατών. Η προστασία των επιβατών ξεκινά, πιστεύω, έχει ως αφετηρία την ενημέρωση, τις πληροφορίες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αναφέρθηκε το ΕΦΣΙ, σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ψηφίωση, ψηφιοποίηση των μεταφορών. Και σε λίγο οι συναδελφοί μου θα σας εξηγήσουν ε, το επόμενο βήμα του CEF, του Connecting Europe Facility και εκεί θα μάθετε πώς χρησιμοποιούμε την δεύτερη, ε, το second call για να βελτιώσουμε τις συνδεσιμότητα μεταφορές. Και τώρα το λόγο έχει και πάλι η συγγητρία για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Για να ολοκληρώσω, αυτό που θα ήθελα εκ νέου να υπογραμμίσω είναι το εξή. Ότι το σημείο αφετηρία είναι ότι οι νέε υπηρεσίε, η δημιουργία είναι αρνητικό στην Ευρώπη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ε, βάσει κοινών και ίσων όρων. Δηλαδή, οι φορείς ε, της αγοράς και οι νέοι φορείς ε, της αγοράς θα πρέπει να ελέγχουν την αγορά. Και από εκεί και πέρα, από πλευρά του ο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι και οι παλιοί και οι καινούργοι φορείς είναι παίζουν με ίσους όρους, ότι δεν υπάρχει ονικό ντάμπινγκ, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή και ότι ε, λειτουργούν όλα αυτά όπως και τα συστήματα μεταφορών για προσαφαλή του πολίτη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τα... την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δεν μπορούμε να παρατείνουμε άλλο περίπτωση της εργασίας μας γιατί θα ψηφίσουμε αύριο στις 9. eigentlich jetzt zum... Θέλαμε να περάσουμε στο πέντε της ημερήσιας διατάξης για την παρουσίαση της Επιτροπής DG Move για το επόμενο πρόγραμμα εργασίας για το Connecting Europe σε ό,τι αφορά την δεύτερη πρόσκληση υποβολής προσφορών. Θα έπρεπε να έχει καταφτάσει στις 4, αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Έχει κάποια εξήγηση να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ja, das, äh, Σας καλωσορίζω λοιπόν στην επιτροπή μας. Κάτι σε 11 λεπτά. Το δεχόμαστε. Αυτό που δεν δεχόμαστε, σας παρακαλώ ακούστε μας με προσοχή, είχατε στις 30, ε, στις 30 Οκτωβρίου για την ε, εφαρμοστική πράξη για την ευκόλυνση και κάνετε μια σχετική ανακοίνωση στον τύπο στι 5 Νοεμβρίου. Και το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για τι 86 αυτές σελίδε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν ε, το δεχόμαστε. Ε, μα, πρώτα ενημερώνετε τον τύπο και μετά το Κοινοβούλιο. Τόσε σελίδε, λοιπόν τι λάβαμε την Παρασκευή και καλούμαστε σήμερα να τη συζητήσουμε. Θυμάστε και τι έγινε στον τριμερή διάλογο που το Συμβούλιο μας ε, έδωσε 70 σελίδες το προηγούμενο βράδυ για να τα συζητήσουμε το επόμενο, την επόμενη μέρα. Απορρίψαμε λοιπόν ε, τη διαδικασία και έκτοτε το Συμβούλιο μας δίνει τι σχετικές τα έγγραφα τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. θα κανουμε μία εξαίρεση σήμερα αλλά τουλάχιστον όταν ενημερώνεται τον τύπο, ενημερώνεται και την κοινοβούλιο. Και σα δίνω λοιπόν το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τα όσα είπατε. Να ζητήσω λοιπόν πρώτα συγγνώμη για αυτό και να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά. Ναι, θα είμαστε ε, πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Θα φροντίζουμε να ενημερώνεστε επαρκώς πριν κάνουμε οποιαδήποτε ανακαίνιση στον τύπο. Εντάξει, δεδομένου αυτό φυσικά αυτό που είναι σημαντικό είναι η ποιότητα της πληροφορία και η πληροφορία που δόθηκε στον τύπο ήταν πάρα πολύ σύντομη. Δεν είχαμε ευκαιρία να εκφραστούμε όπως έχουμε σήμερα εδώ μαζί σας σε αυτή την Επιτροπή και επίση ε, και να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος διμερό ε, στο πλαίσιο κάποιας παρουσίαση. Έχουμε προετοιμάσει μια παρουσίαση για εσά. θα σας την αφήσουμε διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό υλικό το οποίο μπορείτε να διατηρήσετε ως υλικό αναφοράς το οποίο μάλιστα μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να μας υποβάλλετε και περισσότερες ερωτήσεις. Θα περιοριστώ σε κάποιες ε, λίγες σημαντικές πτυχές ε, σε αυτή τη δεύτερη έκκληση για, στο πλαίσιο τη διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη και ελπίζω να προλάβουμε να έχουμε και κάποια συζήτηση σήμερα και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για τεχνικές συναντήσεις ε, αλλά και θεματικές συναντήσεις εφόσον το επιθυμείτε επί συγκεκριμένων ε, θεμάτων. Αυτή είναι η δεύτερη ε, πρόσκληση η υποβολή προσφορών. Η πρώτη ήταν μεγάλη επιτυχία. Ε, υιοθετήσαμε 276 ε, έργα για συνολικό ποσό, ποσό χρηματοδότησης 13,1 δις. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, διότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται τη βοήθειά μας οι δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη και όσοι προωθούν διάφορα προγράμματα ώστε να αποκατασταθούν οι επενδύσεις σε υποδομές και να γίνει καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της διευκόλυνσης. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να συγχαρούμε και εσά για τις σοφές επιλογές που έγιναν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτής της διευκόλυνσης, όχι μόνο όσον αφορά τα χρηματικά ποσά, αλλά και όσον αφορά τις προτεραιότητες. Αποδειχθήκε ότι ήταν σωστές οι επιλογές υπό την έννοια ότι είχαμε πολλά έργα υψηλή ποιότητα, τριπλάσια ζήτηση από ό,τι υπήρχε διαθέσιμο και γι' αυτό το λόγο ένα χρόνο μετά από την πρώτη πρόσκληση υποβολή προσφορών θελήσαμε να βρισκόμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε μια δεύτερη πρόσκληση υποβολή προσφορών η οποία θα χρησιμοποιηθεί από εμά, φυσικά όσο το δυνατόν καλύτερα για να αξιοποιηθούν οι υπόλοιποι οικονομικοί πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, σημαντικό ποσό αποτελείται από δύο μέρη 1,1 δις ε, για όλα τα κράτη-μέλη και 6,5 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα από το Οικονομικό Κονδύλιο των κρατών μελών ε, της πολιτικής συνοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση αυτής της αυτών των προσφορών που θα δοθούν εδώ θα εξετάζει τρεις πτυχές. Πρώτον, ε, την προτεραιότητα, κατά πόσο δηλαδή το εν λόγω έργο αποτελεί προτεραιότητα ή όχι και αυτή τη φορά έχοντας τα εγκεκριμένα σχέδια εργασίας ε, ε, που έχουν εκδοθεί από τους συντονιστές, ε, αυτά τα σχέδια εργασίας θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγή για την αξιολόγηση του βαθμού προτεραιότητας ενός έργου. Δεύτερον, ένα κριτήριο που διατηρείται η οριμότητα του έργου, που θα είναι επίσης αποφασιστικός παράγοντας, και τέλος, τρίτο κριτήριο που είχε χρησιμοποιηθεί και στην προηγούμενη πρόσκληση για υποβολή προσφόρων αλλά αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία αυτή τη φορά επειδή το συνολικό ποσό των κοντιλίων ε, φτάνει ε, έχει σχεδόν εξαντληθεί, φτάνει στο τέλος του, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα ακριβή ποσά χορηγιών που θα ε, απαιτηθούν για συγκεκριμένα έργα ώστε να μεγιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όχι μόνο τα νέα οικονομικά ε, εργαλεία στο πλαίσιο του ΣΕΦ ε, όπου έχουν δεσμευτεί 140 εκατομμύρια ε, ευρώ για αυτά τα μέσα αλλά και να τα αξιοποιήσουμε αφού τα έχουμε πληρώσει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διευκόλυνση αυτή τη συνδέεται στην Ευρώπη, τη διευκόλυνση CEF. Και με χαρά μου έχω να πω σήμερα ότι η συζήτηση και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για όλα αυτά είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Ο Στεφάν έχει αναγραφεί στο Λουξεμβούργο, όπου περνάει τουλάχιστον δύο μέρε τη βδομάδα συνεργαζόμενο με την τράπεζα και σύντομα θα ανακοινώσουμε τα πραγματικά προγράμματα ε, μεταφορών στο πλαίσιο της ε, ΣΥΦ, γιατί πολλά έργα αναφέρονται ως ΣΥΦ, αλλά ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να σας ανακοινώσουμε ε, πραγματικά έργα μεταφορών. στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Το Γενικό Τροκονδύλιο θα δεσμευτεί για βάσει όλων των νέων μέτρων που μας βοηθήσατε να εντάξουμε στον κανονισμό ΣΕΦ πρώτα απ' όλα ε, καινοτομία και νέες τεχνολογίες ε, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και την πρόθεση των εναλλακτικών καυσίμων την αστική διάσταση τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση της σύνδεσης των αστικών κόμβων με το συνολικό δίκτυο ε, θαλάσσιες οδοί όπου αναμένουμε κάποια έργα πολύ ψηλής ποιότητας ε, ε, συνολικά συστήματα διαχείρισης μεταφορών για κάθε είδους μεταφορά και εδώ έχουμε την κλασική γραμμή ITS για τις οδικές μεταφορές το CESAR που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία όλους μας έχει εκπλήξει ψηλή ποιότητα και το πλήθος των έργων που υποβλήθηκαν στην πρώτη πρόσκληση το ITMS ε, μέσω του οποίου διασφαλίσαμε δύο φορές 200 ε, εκατομμύρια για το ITMS ε, και αυτό θα ε, καθοδηγείται από τις κατευθύνες αρχές του τέταρτου πακέτου σιδηροδρόμων και με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς μαζί για, τα, και, για τους οργανισμούς που θα συμμετέχουν και τα River Information Systems, χαμηλό, μικρότερες κλίμακες φυσικά. Όσον αφορά τα κονδύλια, εδώ μας εξέπληξε ε, οι εξαιρετικές ε, προτάσεις στο πλαίσιο των χωρών του, της πολιτικής συνοχής ε, και οι προτάσεις που να Βλέπουμε θετικά τη χρήση του υπολείπου κονδυλίου συνοχής σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προσφορών για δεύτερη φορά φυσικά και πάλι για σημαντικά έργα, για έργα υψηλής που ε, παρατηρούνται στο παραρτημά Μαζί με αυτή την πρόσκληση υποβολής προσφορών ε, θα τρέχουν και άλλες δραστηριότητες για τις νέες ε, χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις. Ε, το ανέφερα πριν από λίγο λεπτά. Και πάλι επαναλαμβάνω είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί στο μέγιστο δυνατό ποσοστό με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από αυτά τα νέα χρηματοοικονομικά συστήματα ε, χρηματοδοτικά συστήματα, συγγνώμη. Το επόμενο βήμα θα είναι η, να ε, διοργανώσει μια ενημερωτική μερίδα που θα αποτελέσει την επίσημη αφιτηρία αυτή τη νέα πρόσκληση, ε, θα λάβει χώρα 30 Νοεμβρίου εδώ στι Βρυξέλλες και θα μα έκανε καλή, μεγάλη χαρά η συμμετοχή κάποιων από εσά σε αυτή την εκδήλωση. Η πρόσκληση υποβολή προσφορών θα είναι ανοιχτή μέχρι μέσα Φεβρουαρίου του 2016. Όπως, λοιπόν και με την πρώτη πρόσκληση θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την επιλογή των έργων στις αρχές του καλοκαιριού του 2016 και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε εδώ να επικοινωνήσουμε μαζί σας αρχές Ιουνίου για να σας παρουσιάσουμε την περιγραφή των τύπων των έργων που θα μπορούσαν να επιλεγούν σε αυτό το στάδιο πριν ουσιαστικά προχωρήσουμε με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των 20 ημερών που θα λάβουν χώρα στο Ρότερνταμ από 20 κάπου από 20 και 22 Ιουνίου. Εύχομαι λοιπόν ότι όπως και τις προηγούμενες φορές ε, θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή ε, ε, ε, των μελών του Κοινοβουλίου στις ημέρες 10 ή 20 με 22 Ιουνίου στο Άμστερνταμ είναι σημαντικό γιατί θα έχουμε και μια διάσκεψη που θα, βασίζεται, που θα αφορά τα εμπορεύματα, τα συνδρομικά εμπορεύματα και ελπίζουμε μεγάλη συμμετοχή από εσάς στη διάρκεια της εκδήλωσης. Αυτά όσον αφορά την εισαγωγή, ε, δεν ακολούθησα την παρουσίαση, δεν χρησιμοποίησα την παρουσίαση για να σας μιλήσω εδώ. Θα σας την αφήσω όμως για να επανελθείτε με ερωτήματα και για να αφήσω και λίγο χρόνο για να μπορέσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ και φυσικά σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και για το κείμενο που μας δώσατε. Το θέμα που μας απασχόλησε ήταν μόνο ε, η χρονική στιγμή. Οι δύο εισηγητές τώρα είναι σαν για Σέντρος και θα έχει το λόγο. Όχι. Οι εισηγητές έχουν πρώτη το λόγο. Εδώ και δεκαετίες, κυρία Αγιάλα Σέντερ. Αν δεν θέλετε, δεν θέλετε. Δεν σας υποχρεώνουμε. <laughs> Okay. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Είχα την εντύπωση ότι το λόγο θα είχαν οι συντονιστέ. Τέλο πάντων. Γι' αυτό είχα ζητήσει από τη γραμματεία να, να με καταχωρήσουν για μετά. Τέλο πάντων. Να ευχαριστήσω το Μισιόν. Είναι αλήθεια ότι πάντα έτσι μας ευνηδιάζουν. Δεν θα έβλεπτε μία ενημέρωση. Εγώ ήμουν ε, ασχολούμαι με τα θέματα θαλασσίων μεταφορών και ευνηδιάστηκα. Καλό θα ήταν, γιατί ξαφνικά είδα ότι θα υπήρχε, θα υπήρχε αυτή η παρουσίαση. Καλό θα ήταν η Κομισιόν τουλάχιστον 12 ώρες πριν να μας αποστέλει μια έκθεση. 10-12 ώρες, τι να πω να μην το βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας γιατί έχουμε και πάρα πολλές εκπροσωπούμε πάρα πολλές περιφέρειες ε, πολύ ευαίσθητες αυτά τα θέματα εν πάση εγώ θα ήθελα να πω απλώς ότι περιμένουμε την ε, μελέτη απάντησης των κρατών μελών που είχαν την γενεοδορία να μας υποβάλουν σε, κοινό, σε κοινή ψήφο τους πόρους ε, συνοχής ε, και με ικανοποιεί το γεγονός ότι ε, καταφέραμε να προβλέψουμε ένα τμήμα της ΕΦΣΗ για πιο οριζόντια θέματα γιατί στους μήνες υλοποίησης που έχουν περάσει ε, υπάρχει πολλή συζήτηση, έχουν ενεργοποιεί διάφορα φόρα, υπάρχουν προτάσεις τροπολογίας για να τις πω έτσι, για να τις πω δηλαδή. Ε, καλό θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουμε και στο τμήμα το πιο ενωσιακό, για να το πω έτσι. Και στο εδαφικό και στο ευρωπαϊκό. Καλό θα ήταν να μας εξηγηθεί λοιπόν κάπως καλύτερα αυτό που είχαμε δει και στην άλλη συνεδρία, στην προηγούμενη συνεδρίαση των περιφερειών σχετικά με το θέμα των διαδρόμων. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού ήμασταν πάρα πολύ εστιασμένοι στο κεντρικό ούτως υπήν τμήμα δηλαδή το ενωσιακό. Η Κομισιόν τώρα μας λέει ότι υπάρχουν διάφορα, διάφορα σημεία συνοστισμού ε, για τις διασυνοριακές ε, κινήσεις κτλ. Αλλά είναι σημαντικό η Κομισιόν να διατηρεί υπόψη της την αναγκαιότητα της πρόβλεψης που είχε τεθεί. Γιατί οι συντονιστές συζητούσαν ε, την τροφοδότηση των διαδρόμων, αλλά εν πάση η ιδέα του δικτύου που ήταν πιο ισορροπημένη και με το ITS, αλλά και εν πάση ε, με ένα πιο οριζόντιο χαρακτήρα, ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση, αντιστάθμιση. Ιδάλλως δίνουμε την εντύπωση ότι θέλουμε να ικανοποιήσουμε και να εξυπηρετήσουμε απόλυτα το κέντρο και την περιφέρεια την ξεχνάμε λίγο. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ε, θα μπορούσαμε να επιλύσουμε κάποιες από αυτές τις επικρίσεις ε, που έχουμε από την περιφέρεια χρησιμοποιώντας πόρους που έχουμε στη θέση μας, αλλά η Κομισιόν καλό θα ήταν ε, να προχωρήσει σε μια πληρέστερη εξήγηση ότι, να μας πείσει δηλαδή, ότι με αυτούς τους διαδρόμους δεν εξυπηρετούμε για μία ακόμα φορά το κέντρο κατά της περιφέρειας. Ενώ η περιφέρεια που ήδη εξυπηρετείται λιγότερο πλήρως για να το πούμε έτσι θα μπορούσε να υποφεληθεί πολύ περισσότερο από αυτές τις ροές. Ευχαριστώ. Danke σας ευχαριστώ. Ντομινί Κρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν για αυτές τις πληροφορίες. Δεν θα επανέλθω στη χρονοδιάγραμμα και στο πώς ε, χειριζόμαστε το κοινοβούλιο που θα πρέπει να το μεταχειριζόμαστε λίγο καλύτερα από τον τύπο. Τέλος πάντων. Έχω πολλές ερωτήσεις και πολλές παρατηρήσεις. Φυσικά χαίρομαι που τηρούμε τα δύο βασικά κριτήρια, το... τη σκοπιμότητα και την οριμότητα των έργων. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας όλο αυτό. Με ενδιαφέρον παρατηρώ ότι αλλάζει η νοοτροπία. Τα οριζόντια έργα γίνονται όλο και πιο σημαντικά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αυτό μεταφράζεται σε μια βελτίωση των συμμετοχής της προσκλήσης υποβολή προσφορών γιατί παλιά όταν μιλούσαμε για το ΣΕΦ νομίζαμε ότι μιλούσαμε για περιφερειακές ε, δραστηριότητες ε, ε, είναι λοιπόν όλο και σημαντικότερα τα οριζόντια σημεία οργάνωση κτλ. Και το πρώτο ερώτημα που έχω προ την Κομισιόν είναι το εξή. Το ζήτημα των χρηματικών μέσων στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility. Γνωρίζουμε ότι στη συζήτηση ε, για το ΕΦΣΥ υπήρξαν ε, διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν ε, για τη δέσμευση ενός κομματιού το οποίο θα μεταφερόταν σε επιχορηγήσεις. Να υπενθυμίσω ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΣΥΕΦ είναι, βρίσκονται σε, ένα, σε μια κοινή δεξαμενή κινδύνου με άλλα μέσα ε, με άλλα ταμεία παρόλα αυτά δεν αλλάζει το είδος, ο τύπος ε, του χρηματοδοτικού μέσου δεν είναι διαφορετικός ε, από του ΕΦΣΥ βασίζεται στην ίδια νοοτροπία και αυτό που δεν καταλαβαίνω θα θέλω να μας εξηγήσει η Κομισιόν είναι το εξή που θα σε, σε ποια περίπτωση θα στρεφόμαστε προς το σχέδιο Juncker και σε ποια ε, περίπτωση προς το Connecting Europe Facility. Μήπως θα ήταν πιο λογικό να μεταφέρουμε το σύνολο των διαθέσιμων ε, σε επιχορηγήσεις. Το λέω παρότι εγώ υπερασπίστηκα θερμά τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού. Ε, το δεύτερο ερώτημα που έχω Όσον αφορά τα ταμεία συνοχής, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο μέρος του μηχανισμού, δηλαδή τα ταμεία συνοχής παραδίδονται στα κράτη-μέλη ε, βάσει του ποσοστού αναλογίας. Ε, ε, ο καταμερισμός αυτός παρουσιάζει δυσκολίες. Η Κομισιόν πώς θα δεσμεύσει τα κονδύλια αυτά. Γιατί δεν μπορεί να βάλει όλα τα ταμεία στο ίδιο σύστημα. Έχει μια αναλογία να τηρήσει. Οπότε κάποιε χώρε μπορεί να έχουν οριμάσει λίγο περισσότερο από άλλε όσον αφορά τα έργα που καταθέτουν. Αυτό δεν θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα καταμερισμού γιατί από το 18 θα έχουμε μια κοινή δεξαμενή. Δεν πρόκειται λοιπόν να εμφανιστούν κάποιε δυσκολίε. Και η τρίτη και τελευταία μου ερώτηση. Παρατηρούμε διάφορε τεκμηριωμένε μελέτε για την καθυστέρηση των επενδύσεων στα κράτη-μέλη τη Ευρώπη και αντιλαμβανόμαστε ότι οι καθυστερήσει αυτέ οι επενδυτικέ. Ε, είναι σημαντικότερες από ό,τι είχε προβλεφθεί με την κρίση του 2008. Δηλαδή στη Γερμανία, όπως ξέρετε, υπάρχουν καθυστερήσεις επένδυσης και τώρα βλέπουμε ξαφνικά νούμερα για τη Γερμανία ε, αρκετά σημαντικά και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα ε, της επικράτειας μαζί και με άλλα κριτήρια βέβαια. Η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να τηρηθεί κάποιο χρόνο. Θεωρεί η Κομισιόν αφού ε, έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες για να συζητήσουμε τα δημοσιονομικά ε, πιστεύετε ότι μπορεί να προβληθεί κάποιος μηχανισμός επαναχρηματιδότησης του ΣΥΕΦ. E ε, υπάρχει τέτοια πρόθεση να τροποποιηθεί λοιπόν ε, ο τρόπος χρηματοδότησης και δεύτερον ε, έχει αρχίσει να σκεφτεί κανείς ε, τι θα γίνει, θα συνεχιστεί, θα επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα. Ενδεχομένω ε, σε κάποιο άλλο οικονομικό πλαίσιο ή χρησιμοποιώντα άλλε διευκολύνσει, άλλα μέσα. Διότι αυτό παρατήρησαν όλοι, ότι από τα 50 δι πέρασαμε σε κάτω από 30 δι διαθέσιμα, τα οποία ουσιαστικά θα αναλωθούν εντό ενό έτου. Και οι ανάγκε που εξέφρασαν τα κράτη-μέλη, άλλοι ε, ενδεχομένως μετέχοντες ε, ήταν, ε, αντισχούσαν σε τριπλάσια, τραπλάσια ποσά από τα διαθέσιμα που είχαμε. Είτε λοιπόν εδώ μιλάμε για έναν εφιάλτη, δηλαδή σας πρότειναν προγράμματα που δεν αξίζουν τίποτα χωρίς τις ανάγκες που αναφέρθηκαν είτε οι ανάγκες είναι τόσο ψηλές όπως δείχνουν και οι μελέτες έλλειψης επενδύσεων οπότε εκεί πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε λοιπόν είναι θα μείνουμε λέγοντας ότι συγγνώμη 30 δις είχαμε και αν θέλουμε περισσότερα ε, και εδώ αναφέρομαι στους μηχανισμούς επιχορήγησης ε, δεν, μην το συγχαίωμα με το σχέδιο Juncker αυτό λοιπόν θα απασχολήσει την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ε, ή μέχρι το 2020 δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα για νέα προγράμματα. Θεωρώ ότι είναι πρωταρχή σημασία ε, αυτό το ερώτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσκλήσει λοιπόν για υποβολέ προσφορών και αυτή τη φορά και την προηγούμενη φορά καταδεικνύουν ε, αυτό που λένε και οι μελέτε έλλειψη επενδύσεων. Ότι είμαστε 5 ή 10 φορέ ε, κάτω από το αναγκαίο. Προτίθε λοιπόν η Κομισιόν να κάνει κάτι ή το αναγκαιο προτιθεται λοιπον η κομισιον να αυτό θα παραμείνει στον τουλάπι για την επόμενη δεκαετία. Κάτι που θα μπορεί να αποδειχθεί καταστρεπτικό και για το σχέδιο και για την οικονομία μας. Ευχαριστώ Μάρκος Πίπερ επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για την πολύ πιστική παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά τα κρατημέλη και όσα μας λένε για την πρώτη, τον πρώτο γύρο υποβολής προσκλήσεων, υποβολή προσφορών, θεωρώ ότι τα πράγματα ήταν πολύ θετικά και ρώτησε ο συνάδελφος τι θα γίνει με το μέλλον του CEF. Θα πρέπει να υπάρχει ίσως λίγο πιο μεγάλη κατανόηση στο Συμβούλιο, ότι δεν είναι όλα αρνητικά τα οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως να μην σκεφτόμαστε μόνο τον τομέα των μεταφορών, αλλά και τα κράτη-μέλη και να βρούμε και να δούμε ότι βρήκαμε μια δίκαιη, ένα δίκαιο σύστημα. Συμφωνήσαμε με δυσκολία τα όσα αφορούν τα κόντυλα συνοχής και υπάρχει μια διαδικασία όπου δέκα δισεκατομμύρια έχουν κορυφθεί στις χώρες συνοχής στις επόμενη, στην επόμενη περίοδο 6,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ πέρα θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς εκτιμά τις δυνατότητες επιτυχίας του διαγωνισμού αυτού. Υπάρχουν στις χώρες σε επαρκή αρκετά ε, ποιοτικά προγράμματα. Οπότε να υπάρχει χρηματοδότηση στον τομέα των μεταφορών ή ενδεχομένω να πρέπει να ψάξουμε να βρούμε δυνατότητες αν δεν ε, το πετύχουμε αυτό στην δεύτερη υποβολή προσφορών. Τα κοντήλια αυτά να χρησιμοποιηθούν σε τομεί που είναι συγγενικοί με τον τομέα μεταφορών, αλλά στι χώρε συνοχή και πάλι. Είχαμε διαπραγματευτεί τότε ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να μείνουν στι χώρε συνοχή. Και θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω από πλευρά τη Επιτροπή Μεταφορών σε αυτό. Αλλά τι σημαίνει αυτό σε σχέση και με την επόμενη περίοδο, το έτσι αυτό Ενρίκε. Θα πρέπει να το σκεφτούμε από τώρα ουσιαστικά το τι θα γίνει σε σχέση με το τη διευκόλυνση αυτή, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και νομίζω ότι η εμπειρία καταδεικνύει και στα κρατημέλη πόσο σημαντικό είναι το μέσο των μεταφορών. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω κατεπηγόντω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα προετοιμάσει αυτά και να δει τι θα κάνει στο μέλλον και να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίζει και να διαφημίζει το Connecting Europe Facility. Να τονίσω ένα τελευταίο θέμα, η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Έχω την εντύπωση ότι κάπως τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Γιατί δεν είναι τόσο σαφή, αν ξέρετε, η σύνδεση στο ΕΦΣΥ, στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων διαγράφεται όλο και πιο έντονα ότι στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουμε πραγματικά εξαιρετικά προγράμματα. Αλλά αν τα καταφέρουμε θα έχουμε και μια χρηματοδότηση η οποία θα καλύπτει όλους τους τομείς της, ε, των μεταφορών. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο πιο προς το συμφέρον το ιδιωτικό θα συνδεθούν με τους σιδηροδρόμους, με τις ε, οδικές μεταφορές και έτσι λοιπόν ενδεχομένως θα υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή από πλευρά των ιδιωτικών επενδυτών, για παράδειγμα το τούνελ στη Μπρέμεν. Θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται με τέτοιο τρόπο προκειμένου να υπάρχει ε, διπλή ε, επιδότηση και για τις οδικές μεταφορές σε ό,τι αφορά δηλαδή τα δύο που θα ζητούνται και σε ό,τι αφορά τη συνδρομική μεταφορά. Δηλαδή, να υπάρχει όρος συγχρηματοδότησης και συγκεκριμένων διαδρόμων. Ίσως να γελάει ο Ντόμινικ. Έτσι λοιπόν, με την εξισορρόπηση των κινδύνων, να σπρώξουμε και τους ιδιωτικούς επενδυτές προς επενδύσεις οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο δυναμικό θα παρακαλούσα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί προ την κατεύθυνση αυτή. Επόμενο ομιλητή. Θα είμαι σύντομη, λέει η κυρία Μάιστερ, γιατί πολλά από αυτά που με ενδιαφέρουν ε, τα θέσατε ήδη. Αυτά που είπε ο Ντομινίκ, θέλουμε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρω το χωρί να πάνε πράγματα και κονδύλια από το ΕΦΣΥ στο θέμα αυτό. Και ο Μαρκούς Πίπερ ανέφερε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τους συνδεδρόμους, τις πλευρές μεταφορές και επίσης με απασχολεί το θέμα των χωρών συνοχής. Θα πρέπει να δαπανώνται τα κονδύλια με σκόπιμο και σωστό τρόπο. Και έχω και άλλη μια ερώτηση η πρώτη δόση δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη όλα αυτά που ζητήθηκαν. Δεν ανταποκριθήκαμε δηλαδή σε όλα τα αιτήματα. Υπάρχει κάποια διαδικασία ώστε τα έργα αυτά που δεν χρηματοδοτήθηκαν στην πρώτη δόση να είναι στην κορυφή της λίστας τώρα. Και μετά, λέει ο πρόεδρος, θα πάρω και εγώ το λόγο. Η πρόταση αυτή ήταν πάρα πολύ καλή σε ό,τι αφορά τον διεθνωριακό κλάδο. Είχαμε για παράδειγμα τα πρώτα τα μεγάλα προγράμματα και μετά τα μικρότερα προγράμματα. Λιόν Τουρίνο. 12, 14 δισεκατομμύρια. Κανένα πρόβλημα. Αλλά 102 εκατομμύρια για ένα μικρό πρόγραμμα τελικά φαίνεται ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Να υπάρχει λοιπόν ένα συνδυασμό να δίδονται και μεγάλες ε, επενδύσεις για μεγάλα προγράμματα, αλλά σε συνδυασμό με δύο-τρία μικρά. Δεύτερο ερώτημα για την Κροατία. Ακούσαμε ότι η κροατική κυβέρνηση για τον Τράμπα ε, ζήτησε τρία α, υδροελεκτρικά αεργά. Η Τράμπα είναι ο Αμαζόνιος ε, της Ευρώπης. Και δεν έλαβαν στην πρώτη δόση καθόλου χρήματα, κανένα κοντέλιο. Και να είστε σίγουροι ότι δεν του άρεσε και ιδιαίτερα. Οι κυβερνήσει τώρα λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να το ξαναθέσει το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι λόγοι, οικολογικοί και το καθεξής. Αλλά μπορεί να θέσει αυτό το πρόγραμμα εκ νέου η κυβέρνηση ως υποψήφιο. Μπορεί, το έκανε και ποια θα είναι η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τώρα λοιπόν σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Thank you. Ευχαριστώ. Και πάλι ζητώ συγγνώμη για το ευνίδιο της παρουσίας αυτής. Είχαμε προσπαθήσει να έχουμε νωρίτερα, είχαμε ζητήσει. Εν πάση θα προσέξουμε την επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα. Λοιπόν, Νομίζω ότι υπήρξε μια κάποια σύγχυση με την μεταφορά των πόρων στο έύση των πόρων συνοχής. Διότι δεν επελέγησαν όλα τα έργα. Το οποίο σημαίνει ότι τα είχαμε εξετάσει προσεκτικά τα έργα αυτά. Τώρα μας ρωτάτε, ήσασταν εξίσου αυστηροί με τα έργα συνοχής όπως και με τα άλλα. Ναι, η απάντηση είναι οπωσδήποτε ναι. Ωστόσο βλέπουμε ότι η ποιότητα των έργων είναι εμφανή τουλάχιστον εκείνων που έχουν επιλεγεί στην πρώτη κλίση. Και στη δεύτερη κλίση θα χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των εθνικών φακέλων. Δηλαδή, δεν θα έχουμε το θέμα του να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να στηρίξουμε με άλλους πόρους. Και βεβαίω παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δεύτερης κλίσης ΕΦΣΥ, που θα τα συζητήσουμε μαζί σας, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι σε εθνικούς φακέλους, θα δούμε αν μπορέσουμε να διοργανώσουμε και μια τρίτη εκτακτή κλίση, έκτακτο διαγωνισμό. Όμως, βεβαιώνω ότι τα έργα είναι υψηλής ποιότητος διότι οι οργανωτές τους συνεργάζονται ενεργά με την ίνεα τον οργανισμό που έχουμε συστήσει για να προετοιμάζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του φακέλου αυτού κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καθότι έχουμε μια καινοτόμα προσέγγιση, έχουμε όλοι συμφέρον να δείξουμε ότι αυτό λειτουργεί και ότι επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μεγαλύτερο ποσοστό την μεταφορά ή το εύση της πολιτικής συνοχής. Και η ανταπόκριση από τα κράτη συνοχής είναι εξαιρετική. Θεωρούν ότι η ευκαιρία αυτή είναι πολύ χρήσιμη, πολύτιμη και βλέπουν επίσης ότι ως προς το χρονοδιάγραμμα μπορούμε να τους βοηθήσουμε με την υλοποίηση των έργων αυτών πολύ ταχύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε μέσω άλλων μέσων. Εξού και το 6,5 δις που είναι το υπόλοιπο του φακέλου συνοχής, ότι μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας έργα στη δεύτερη κλίση. Οριζόντια θέματα τώρα. μία δική σας κριτική που λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη και δεν ήταν έκπληξη γιατί το παράρτημα του κανονισμού εύση είναι σαφέστατος αλλά είδαμε ότι πολλοί πόροι είχαν δεσμευτεί από μεγάλης κλίμακας έργα στην πρώτη και, στην κλίση, και όχι αναγκαστικά μεγάλα έργα στην περιφέρεια όπως είπατε κάποιοι από εσάς και γι' αυτό κάναμε την επιλογή να προσπαθήσουμε να εστιαστούμε επί οριζοντίων θεμάτων για να έχουμε καλύτερη ισορροπία και να έχουμε και μέτρα χρηματοδότησης που να προωθούν την αποτελεσματικότητα όλου του δικτύου. Τώρα, το να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις επιλογής, αν θέλετε, μεταξύ μεγάλων ή μικρών έργων, αυτό είναι ένα κριτήριο που δεν είναι γραπτό. Το έχουμε στην εσωτερική αξιολόγηση των έργων της ε, πρώτης κλήσης. Και καθότι ήταν τόσο μεγάλο ο αντίκτυπος ο δημοσιονομικό των μεγάλων αυτών έργων, θα μπορούσαν πιο εύκολα να συνδεθούν με μικρότερη κλίμακα έργα. Και έχουμε και την εμπειρία που συλλέγουμε αξιολογώντας αυτά τα έργα στο μέλλον. Θα μπορούσαμε δηλαδή αυτές τις προϋποθέσεις να τις κάναμε ακόμα πιο ρητές. Τώρα, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα εντό του ΕΦΣΥ και η συμπληρωματικότητα με το Ταμείο Juncker Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι καλή η ερώτηση. Με τη δεύτερη δέσμη των 70 εκατομμυρίων, λέει ο μιλτής, μπορούμε περαιτέρω να δείξουμε ότι τα έργα του Ταμείου Συνοχής έχουν μεγαλύτερη αξία στο σύνολο του ΕΦΣΗ. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, να ε, εξωθήσουμε την Τράπεζα Επενδύσεων να πάει προς έργα υψηλότερου κινδύνου, ψηλότερου ρίσκου. Παρότι το σχέδιο Juncker είναι εκεί για να υποστηρίξει σχέδια υψηλότερου κινδύν, επενδυτικού κινδύνου, θα πρέπει να λάβουμε έργα σε ένα λογικό πλαίσιο, εντός λογικών ορίων κινδύνου. Και επομένως θα μπορέσουμε να πάμε στην στη δεύτερη κλίση με υψηλότερο κινδύνου έργα και κυρίως έργα που να συνδέονται με συγκεκριμένες θεματικές. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα έχουμε ένα ταμείο που θα μπορεί να χρηματοδοτείται από το ΣΕΦ και το ERTMS Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε μια πρώτη δέσμη θεματική για, μεταξύ άλλων, το greening, το πρασίνισμα των σκαφών. Για να επικαιροποιήσουμε τον θαλάσσιο στόχο ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί με λιγότερο επιμολυντικές ε, μηχανές και εξαρτήματα. Και στα πλαίσια των μέσων αυτών που θα ήταν καθαρά εντός του ΣΕΦ θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα ταμείο που να είναι απολύτως αφιερωμένο στην ευφυή, στις αφιείς αστικές μεταφορές και στις πιο περιβαλλοντικές δηλαδή. Τώρα μια ερώτηση θα τεθεί όπως είπατε και εσείς και θα τεθεί σίγουρα στα πλαίσια της δεύτερης κλίσης. Τι θα κάνουμε με τους υπόλοιπους πόρους που είχαν δεσμευθεί για τα χρηματοδοτικά μέσα του ΣΕΦ. Θα μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των ταμείων αυτών ώστε να μετακινηθούν προς τις παραδοσιακές χορηγήσεις για να έχουμε και μια μεγαλύτερη κλιμακασή δυνατών τρίτη κλίση του ΣΕΦ για να πάμε και σε πιο παραδοσιακές μορφές επένδυση, αν το πω έτσι. Και για τις καθυστερήσει των επενδύσεων και τις επιπτώσει τους, εκεί πράγματι έχουμε ένα φόρτο εργασία. Σε έργα ε, υποδομών μεταφορών σε όλη την Ευρώπη και το έχουμε καλύψει με διάφορους τρόπους. Το Ταμείο Γιούνκερ ήταν μία από τι απαντήσει, αλλά δεν θα ήταν η μαγική συνταγή για όλα τα προβλήματα. Ήταν ένα από του τρόπους που είχαμε στη διάθεσή μα να ανταποκριθούμε. Άλλος ένας ήταν να τοποθετήσουμε τη χρηματοδότηση των υποδομών σε πιο υψηλή προτεραιότητα πολιτική αν θέλετε. Τρει προεδρίες συνεχής τώρα έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους στο θέμα της χρηματοδότησης υποδομών και εξετάζουμε και διάφορα αριθμιστικά εμπόδια προκειμένου να βοηθηθούμε ακόμα περισσότερο. Όμω, ο ίδιο ο φόρτο εργασία ω τέτοιο. δεν προβλέπουμε ότι θα έχει επιπτώσεις επικαθυστερήσεων έργων που έχουν επιλεγεί υπό το ΣΕΦ. Αυτά που έχουν επιλεγεί υπό την πρώτη κλίση και αυτά που θα επιλεγούν υπό την δεύτερη κλίση, βλέποντας το χρονοδιάγραμμά τους, εκεί βλέπουμε και τον κίνδυνο καθυστέρησης χρονικής. Βεβαίως ο οργανισμός εξακολουθεί να είναι να επιτηρεί όσο μπορεί, και, να, και προσπαθούμε να ελέγχουμε ζωντανά, για να το πούμε έτσι, την ε, ροή των έργων για να αποφύγουμε αυτό το use it or lose it και να έχουμε ανα, ανακυκλωμένους πόρους χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να πάμε σε μια τρίτη κλίση που θα έχει και την παραδοσιακή πτυχή των επιχορηγήσεων. Τώρα, έργα ΕΦΣΙ. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Έργο ΕΦΣΙ καταρχάς δεν σημαίνει οδικού δικτύου αναγκαστικός. Γνωρίζουμε βέβαια, ότι αυτά είναι ευκολότερα και πιο ελκυστικά για τους ιδιωτικούς επενδυτές, χαμηλότερου κινδύνου τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, αλλά τουλάχιστον έχουμε και μη οδικά δίκτυα υπό το εσωτερικές υδάτινες οδείς, το, ο λιμένας του Καλέ, ή έργο που θα χρησιμεύσει για την επαναχρηματοδότηση του Rolling Stocks του σιδηροδρόμους όπως και Περιφερειακό Ταμείο ώστε να χρηματοδοτούνται έργα των αστικών μεταφορών. Τώρα, μπορούν να επανυποβληθούν έργα που δεν είχαν γνωρίσει επιτυχία στην πρώτη κλίση. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει αυτοματισμός και οπωσδήποτε δεν θα ενθαρρύναμε τα κράτη-μέλη να επανυποβάλλουν έργα που δεν έχουν αξιολογηθεί θετικά. Κάτι τη διακοπή λοιπόν μετά τον πρώτο γύρο, εάν είδαμε ότι η δεν επελέγει το έργο επειδή δεν είχαμε τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, τότε υπάρχουν πολύ υψηλέ πιθανότητε να επιλεγεί στη δεύτερη κλίση, στο δεύτερο γύρο το έργο. Αλλά αν δεν έχει αξιολογηθεί θετικά υπό την έννοια των προτεραιοτήτων και τη χρησιμότητό του, τότε προφανώ αυτό δεν θα ήταν αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων σας να επανυποβληθεί, των κρατών μελών δηλαδή. Επίσης θα έπρεπε να δίνετε περισσότερη προσοχή μεταξύ του, του κέντρου, του πυρήνα του δικτύου και του υπολείπου δικτύου. Αυτό που χαρακτηρίσατε κάποιοι από εσά ως ε, περιφερειακό δίκτυο ή καπιλάρι εμπασετώσει. Διακλαδώσεις. Είχαμε ζητήσει από τους συντονιστές να μην εστιάζονται μόνο το κεντρικό κομμάτι του δικτύου, αλλά να βλέπουν και τις υπόλοιπες υποδομές που τελικά είναι ζωτική σημασία προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του core network. Επομένως, κάποιο τμήμα χρηματοδότησης προφανώς θα τοποθετηθεί μεταξύ του core network και του capillary. Τώρα το έργο στο οποίο αναφερθήκατε εγώ δεν το γνωρίζω έτσι όπως το περιγράψατε δεν μου φάνηκε ότι θα ήταν έργο επιλέξιμο υπό την δεύτερη κλίση με την επιφύλαξη του να το ελέγξω καλύτερα το λέω αυτό αλλά δεν έχω ενημερωθεί για κάποιο κροατικό έργο που δεν θα είχε επιλεγεί λόγω κενών χρηματοδότησης. Μάλλον, μάλλον αξιολογήθηκε έτσι αρνητικά. Σας ευχαριστώ και έτσι λοιπόν ε, ολοκληρώσαμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη και περνάμε στη συνάντηση των συντονιστών και θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όσους να από την αίθουσα και τα λέμε αύριο στις 9.